η Γαλλία επλήγει με τον πλέον βίαιο τρόπο. Οι τρομοκράτες ε, επιτέθηκαν με πρωτόγνωρο τρόπο και πρωτόγνωρη ομότητα και βιαιότητα και δολοφόνησαν νέους ανθρώπους, άντρες και γυναίκες, νέα παιδιά. Αυτό το έπραξαν με κτηνώδη τρόπο. Σήμερα λοιπόν ως ε, θεσμός που έχουμε την έδρα μας ε, στη Γαλλία. Για πρώτη φορά μετά την επίθεση βρισκόμαστε σε γαλλικό έδαφος. Γι' αυτό, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω όλους σας για τη συμμετοχή σας ε, στα, ε, στις εκδηλώσεις συμπάθειας, στα συλληπιτήρια που εκφράσαμε στο γαλλικό έθνος, στη γαλλική κυβέρνηση. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ γι' αυτό. Και ε, βεβαίως ε, οι σκέψεις όλων μας είναι στις οικογένειες, ε, τρέφουμε ελπίδες για αυτούς τους βαριά τραυματισμένους να αποκατασταθούν το ταχύτερο δυνατόν. Το ίδιο ισχύει και για τα θύματα του Μπαμάκο και για τα θύματα σε άλλες περιοχές του κόσμου όπου αθώοι άνθρωποι δέχονται επιθέσεις, σφαγιάζονται κατά λέξη από δειλούς τρομοκράτες. Κυρίες και κύριοι, ζούμε σε μια εποχή πολύ μεγάλων προκλήσεων. Ο αριθμός των επιθέσεων, τα οποία, τις οποίες μάλλον οφείλουμε να αναφέρουμε εδώ, γιατί δεν μπορούμε να ιεραρχήσουμε τα θύματα, Κάθε ένα μεμονωμένο θύμα έχει την ίδια ακριβώ αξία για μας. Ο κατάλογος λοιπόν των θυμάτων είναι μακροσκελέστατος. Γι' αυτό τα θύματα του Παρισιού, τα θύματα του Μπαμάκο, όλα αυτά τα θύματα αξίζουν τις σκέψεις μας για τους αθώους σε όλα τα μέρη του κόσμου, στη Συρία, στο Ιράκ, όπου το αυτοαποκαλούμενο Ισλαμικό κράτος έχει παραβιάσει και καταπατήσει όλα τα θεμελιώδη δικαιώματα και αυτό το έχει πράξει με ιδιαίτερη βιαιότητα. Οι σκέψεις ε, λοιπόν ε, στα θύματα μας οδηγούν και σε σκέψεις για τις βίες αυτές πράξεις και αυτά δεν αφορούν μόνο τα θύματα του Παρισιού και του Μπαμάκο και προς τιμήν όλων αυτών των θυμάτων παρακαλώ να γερθείτε από τις θέσεις σας. vielen σας ευχαριστώ πολύ. κυρίες και κύριοι Σήμερα το πρωί είχα το πολύ θλιβερό καθήκον ως ε, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμμετάσχω στο μνημόσυνο του πρώην καγκελάριου της ε, Γερμανίας, του κυρίου Helmut Σμιτ. Με τον Helmut Σμιτ ε, χάσαμε έναν προβεβλημένο πολιτικό, όχι μόνο της Γερμανίας, αλλά της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικά. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, ο κύριος πρώην καγκελάριο Χέλμουτ Σμιτ από κοινού με τον Βαλερή Ζισκάντεστα. Ήταν ένα από τους ιδρυτέ του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματο. Ο Σμιτ όταν ήταν καγκελάριο, αλλά αργότερα και όταν ασχολήθηκε με τα μέσα ενημέρωση, συνέβαλε τα μάλα στην Ευρωπαϊκή Ενοποίηση και στη συνεργασία των λαών πέρα από τα σύνορα. Ο Χέλμουτ Σμιτ, κυρίες και κύριοι, ήταν αρχηγός μιας κυβέρνησης η οποία στη χώρα από την οποία προέρχομαι εγώ βίωσε και αυτή μεγάλη τρομοκρατική απειλή και διαφύλαξε μια αρχή την οποία οφείλουμε και εμείς να διαφυλάξουμε σήμερα. Και αυτό το έχει πει με τα καλύτερα λόγια ο Αλμπέρ Καμού και παραθέτω. Εκείνοι οι οποίοι αποτυγχάνουν στην συμφιλίωση της ασφάλειας και της ελευθερίας αποτυγχάνουν στα πάντα. Αυτά ήταν τα λόγια του Καμού και νομίζω ότι θα πρέπει να τα έχουμε πάντα κατά νου. Αυτό θα πρέπει να είναι το οδηγό νήμα στις πράξεις μας από εδώ και εντεύθεν. Θα πρέπει λοιπόν ε, να ε, διαφυλάσσουμε την ε, ασφάλεια των πολιτών μας και δεν πρέπει ποτέ να επιτρέψουμε εκείνοι που θέλουν να μας τρομοκρατήσουν να καταστρέψουν και τα δικαιώματά μας ελευθερίας. Αυτό είναι καθήκον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κυρίες και κύριοι, τα πρακτικά